Ευρωπαϊκή Ένωση σταδιακά να κινείται και σε όλα τα επίπεδα για να φτάσει σε μια πιο δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαϊφή. Για 4,5 λεπτά ο κύριος Λουίζαντο, Γιάννη Ζαντο, συγγνώμη.